micro is on. Okay. Colleagues, good afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σε ένα λεπτό θα αρχίσουμε, γι' αυτό παρακαλώ καθίστε. Please feel comfortable, take seat. Βολευτείτε και καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας.